Είσουμε ε, ε, ε, αναμένες τις ιδέες του Ζαν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν. Ο κύριος Ριμπέρου Κάστρο για διαδικαστικό θέμα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να προσθέσω τα δικά μου